Good afternoon, uh, everybody. Uh, Χαίρετε. Καλωσορίσατε όλοι στην κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και της Επιτροπής Μεταφορών, ΙΜΚΟ και ΤΡΑΝ αντίστοιχα. Καλωσορίζω τα μέλη και των δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών. Και όπως σας είπα, είναι κοινή η συνεδρίασή μας σύμφωνα με το άρθρο 55 του κανονισμού μας Θα έχουμε κάθε φορά χωριστή ημερήσια διάταξη για όλες τις κοινές μας συνεδριάσεις στο μέλλον και θα έχουμε πάντα συμπροεδρία των δύο προέδρων ή αντιπροέδρων. Θα δώσω το λόγο στον συμπρόεδρό μου τώρα για να κάνει κάποια εισαγωγικά σχόλια για να μπούμε στην ουσία στη συνέχεια. Bien, Μιλήσω γαλλικά. Καλημέρα σε όλους. Όπως ε, το είπε η κυρία Βαν Μποσφουίτ, είναι μια κοινή ε, συνεδρίαση αφού η Επιτροπή ΙΜΚΟ θέλησε να παρέμβει σχετικά με το θέμα αυτό ε, η βάση του άρθρου 55, δηλαδή είναι μια μεικτή εργασία των δύο επιτροπών και η σύνθεση ε, που εργαζόμαστε σήμερα θα είναι η συνήθι σύνθεση για το φάκελο αυτό, για το θέμα αυτό. Δηλαδή με ε, μεικτή συνεδρίαση. Βεβαίως ο φάκελος αυτός ε, αποτελεί αντικείμενο κατανομής, θα ξαναμιλήσουμε, αποτέλεσε και το αντικείμενο ενό μικρού ελιγμού της Επιτροπής ε, για τον οποίο θα δώσει ε, εξηγήσεις. Έχουμε μόνο μία ώρα, προτείνω λοιπόν στην συμπρόεδρο που είναι ταυτόχρονα και συνεισηγήτρια να λάβει τον λόγο ως εισηγήτρια για το θέμα αυτό, εξ ονόματος της Επίτροπης ΙΜΚΟ. Έχετε το λόγο, αγαπητοί Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τώρα θα μιλήσω ως εισηγήτρια στα Ολλανδικά. Έχω τη συνήθεια να μιλάω τη μητρική μου γλώσσα όταν είμαι εισηγήτρια. Πρέπει να σας πω ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματικά ανησυχούμε βαθύτατα για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χειρίστηκε την έκθεση. Δεν έχετε διερμηνία. Πώς είναι δυνατόν. Στα αγγλικά. Στα αγγλικά. Στις άλλες γλώσσες είναι εντάξει. Τώρα, ωραία. Ωραία. Τέλε. Ευχαριστώ, Τζάκι. Ε, έλεγα λοιπόν και το επαναλαμβάνω ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανησυχούμε βαθύτατα για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη συγκεκριμένη έκθεση. Ε, από τους συναδέλφους στο Συμβούλιο μάθαμε ότι δεν υπήρξε ενθουσιασμός από τα κράτη-μέλη, το ξέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό. Επίσης μάθαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προτίθεται να αποσύρει την πρότασή της, αλλά θέλει σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των κρατών μελών να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες και τα προβλήματα. Και όλα αυτά είναι λιμένη απόφαση. Πριν ε, αρχίσουμε καν τη δουλειά μας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θυμίζω ότι παραμένουμε συνομοθέτες. Άρα ανησυχούμε πάρα πολύ και μας λείβει όλη αυτή η διαδικασία. Γι' αυτό θα ήθελα να έχω περισσότερη πληροφόρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για την κριτική του Συμβουλίου, τι τους ενοχλεί και τι ε, πρόκειται να κάνει συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς βλέπει δε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί μας έχετε παραγωνίσει, ε, κανονικά μας αφορά το θέμα. Επίσης έμαθα ότι ε, εσείς απλώς αναδιατυπώνετε κάποιες λεπτομέρειες και δεν έχετε μπει στην ουσία της πρότασης. Μα δεδομένης της απροθυμίας του Συμβουλίου και της αρνητικής υποδοχής Μήπως θα πρέπει να ξαναδείτε όλη την πρόταση. Πόσο μάλλον που ε, είναι πολύ συγκεκριμένο ε, να υπάρχει μια βελτίωση της νομοθεσίας, όχι μια απλή αναθεώρηση. Είναι κρίσιμο αυτό το θέμα. Άρα, τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξετάζεται το ενδεχόμενο να αποσύρετε την σύνολη πρόταση και να κάνετε καινούρια. Εκτός αυτού, ε, έχω και κάποιες παρατηρήσεις και ερωτήσεις επί της ουσίας. Θέλετε ένα εναρμονισμένο σύστημα πιστοποίησης του εξοπλισμού ελέγχου προστασίας των αερομεταφορών ε, και στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς αλλά οι κανόνες έχουν νόημα εφόσον βελτιώνουν την υφιστάμενη κατάσταση, για να υπάρχει και μία προστιθέμενη αξία. Από ό,τι φαίνεται, είναι όλα τα κράτη-μέλη αντίθετα, οπότε θα πρέπει να αναρωτηθούμε, κάτι τρέχει εδώ. Ε, ε, είμαστε σε σωστό δρόμο με αυτή την πρόταση. Και στα πλαίσια της έκθεσης ε, έχω κάνει κι εγώ κάποιες αναζητήσεις και κάποιες μελέτες Υπάρχει προθυμία ε, να προχωρήσει το κράτη-μέλη βάσει ε, των προτύπων ΕΚΑΚ ή e CAC. Και γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί το νέο εναρμονισμένο σύστημα τόσο απαραίτητο και τόσο αναγκαίο. Αυτά είχα να πω στη συγκήτρια και θέλω να δώσω το λόγο ε, στον εισηγητή της Επιτροπής Μεταφορών και δεν έχω το όνομά του εδώ. Ποιος είναι ο κύριος Ντεγκράντες. Α, ναι, είναι ο κύριος Δεγκράντες Πασκουάλ, ε, κύριος Ρικέ, ο οποίος θα λάβει το λόγο ως συνεισηγητής εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και Πρόεδρε και συνεισηγήτρια, εγώ είμαι. μου φαίνεται σπουδαία ιδέα να το συζητήσουμε σε κοινή συνεδρίαση, το, ε, οι δύο επιτροπές Τραν και ΙΜΚΟ και να αρχίσουμε επιτέλους ή δυνατόν να δουλεύουμε, γιατί είναι σκάνδαλο αυτό που συνέβη με τον τρόπο που συνέβησαν. Χάσαμε τόσο χρόνο, γεμάτο αβεβαιότητες, ανασφάλειες. Αυτό είναι το, το πιο βλαβερό που μπορεί να συμβεί στις αερομεταφορές και σε συστήματα ασφαλείας. Επιτέλους ασχολούμαστε με αυτό το θέμα, με την αυστηρότητα που του αρμόζει. Το σύστημα πιστοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον εξαπλισμό ελέγχου προστασίας των αερομεταφορών βρισκόταν έτσι κάπως μετέωρο πολιτικά, για να το πω έτσι, και δύσκολο να το εξηγήσουμε, γιατί ήταν σε αυτό το κενό. Και ομολογώ, όταν με ρωτούσαν τι συνέβαινε, δυσκολευόμουν να εξηγήσω, γιατί συνήθως ήμουν εισηγητή για τους σαρωτές, τους σκάνερ ασφαλείας, που εδώ στο Κοινοβούλιο κάναμε μακρά συζήτηση και βγάλαμε και συμπεράσματα, σωστά. Και τα αφήσαμε όλα στον αέρα. Έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να λάβουν ενδεχομένω αποφάσεις αποφάσει του. Τώρα όμως που αναπόκειται στα κράτη-μέλη να πάρουν ε, υπεύθυνε αποφάσεις για να εγγυηθούν την ασφάλεια, Και η ασφάλεια είναι και αυτή θεμελιώδης δικαίωμα και ε, οι πολίτες το διεκδικούν δυστυχώς αυτό το θλιβερό κόσμο που ζούμε για του γνωστού λόγου, να έχουν δικαίωμα στην ασφάλεια παραπάνω από την ελευθερία. Το Σεπτέμβριο ε, συζητήθηκε και ποτέ στο Κοινοβούλιο, σε κανένα τριμερή διάλογο δεν συμμετείχε το Κοινοβούλιο. Για ποιο λόγο αυτό είναι ανεξήγητο. Να μην σα πω ότι είναι και προσβλητικό σχεδόν. Δεν μπορεί το Κοινοβούλιο να το δεχτεί αυτό, να το επιτρέψει. Μπορεί να υπάρχουν λόγοι για αναβολή, χρονοτριβή, διάλογο μόνιμο με τα κράτη-μέλη που, που διαφωνούν, εντάξει, συνέβη αυτό, αλλά το κοινοβούλιο παραγωνισμένο, το να ενημερώνεται το κοινοβούλιο είναι εκ των όνου κάλεφ. Εδώ τίθεται σε θέμα σεβασμού, θεσμικού. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Από την άλλη, ε, πρέπει να πω ότι η κυρία ε, είχε την ε, ε, ευγενή καλοσύνη να με ενημερώσει και ευχαριστώ γιατί χρειάστηκε αυτό. Εμείς κάναμε και ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας δώσει εξηγήσεις. Εδώ θα μιλήσουμε για τα εμπόδια που γνώρισε η έκθεση από την αρχή. Και ήταν <laughs> λεξικολογικές οι αλλαγές που κάνανε και προτείναν και όχι ουσίες. Ξέρω εγώ, διατύπωσης αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι οι εγωισμοί, οι εθνικοί που δεν θέλουν να επενδύσουν στην ασφάλεια και μέχρι οι αερολιμένες οι ίδιοι που προσπαθούν να και προτιμούν να βάζουν μαγαζιά παρά συστήματα ασφαλείας. Μέχρι και σούπερ μάρκετ έχουν στα αεροδρόμια. Τι να κάνουμε, τα έχουμε συνηθίσει αυτά. Αμφισβητείται ακόμα και η αρμοδιότητα ΕΚΑΚ εδώ. Ορισμένα κράτη-μέλη αναφέρθηκαν και στον κανονισμό 300 2008 για την ασφάλεια. Όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να διευκρινιστούν από Κομισιόν και Συμβούλιο. Ούτε το άρθρο 4 είναι σαφές, γιατί ζητεί από τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν επιπλέον μέτρα ασφαλείας. Αυτό είναι ένας μόνο από τους λόγους ε, για τον οποίο αντιτίθεται το Συμβούλιο. Ή τουλάχιστον έτσι προσπάθησε να δικαιολογήσει την παράλυση στην οποία έχουμε οδηγηθεί. Τώρα θα σας πω ένα προσωπικό σχόλιο ω είναι σοβαρή αυτή η πρόταση, απαραίτητη, έχει προστιθέμενη αξία για τα κρατημέλη, οι έλεγχοι ασφαλείας να έχουν πιστοποίηση και πρότυπα. Κατά την άποψή μου, σήμερα περισσότερο παρά ποτέ, σε αυτά τα, ε, τους καιρούς που ζούμε ε, σαν θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ακριβώς την προστασία και την ασφάλεια των χιλιάδων ε, Ευρωπαίων που κάθε μέρα ταξιδεύουν στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Και αυτό θα είναι και προς όφελος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας Δηλαδή, εμεί συνεχώ επικρίνουμε ε, τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά χάνουμε το τρένο τη τεχνολογία απέναντι στι ΗΠΑ και κινδυνεύουν να μείνουμε εκτό ανταγωνισμού. Άρα είναι πολύ σημαντική η ιδέα αυτή και θα πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει η ευρωπαϊκή πιστοποίηση. Η αερια ε, η ασφάλεια θα πρέπει να είναι προτεραιότητα. Τελειώνω, Πρόεδρε. Ζητώ από το Συμβούλιο να σταματήσει να ε, ορθώνει εμπόδια σε αυτή τη διαπραγμάτευση ή να μα εξηγήσει γιατί έχουμε δοχηθεί σε αυτή την παράλυση. Γιατί δεν υποχωρεί ούτε σπιθαμή. Γιατί δεν μα έχει καλέσει να συναντηθούμε. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει με τρόπο συνετό και λογικό να μας παρουσιάσει μια νέα πρόταση σε σχέση με εκείνη του Σεπτεμβρίου, η οποία φαίνεται να μην είναι ικανοποιητική ως προς τους ορισμούς, το πεδίο εφαρμογή κτλ. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει επιτέλους στο τι συμβαίνει και τι θέλει στο κάτω-κάτω. να έχουμε μια λέσχη συζητήσεων, οι δύο επιτροπές, Τραν και Ίμκο, και να συζητάμε ε, φιλολογικά, φιλοσοφικά ή να κάνουμε διδακτορικά. Τι θέλει η Επιτροπή, να σας πω τι θέλω εγώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεδομένης κατάστασης να αποσύρει την πρότασή της και δεν είναι νομολόγητο αυτό, ούτε χρειάζεται να ντρέπεται κανείς. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα. Να αποσύρει την ε, πρόταση αυτή και να δεσμευτεί, να κατεβάσει καινούρια με τις γραμμές που έχουν ε, ορίσει ενδιαφερόμενοι. Και γρήγορα. Τώρα να συζητήσουμε θεωρητικά ένα κείμενο που ούτε κατά διάνοια δεν ήταν συνενετικό στο Συμβούλιο και, και οι επιτροπές μας είναι δεμένες χειροπόδαρα και πιστάγωνα, τι να το κάνουμε. Εδώ είναι θέμα συναπόφασης. Ε, αφού βλέπετε ότι το Συμβούλιο αποκλείται να συμφωνήσει, αποσύρετε την πρόταση και βοηθήστε και τις δύο επιτροπές μας που θα πρέπει να συνεργαστούν για να προχωρήσουμε ε, αυτή την υπόθεση. Αυτά προς το παρόν, τίποτα άλλο, κυρία Πρόεδρε και κύριε Πρόεδρε και σταματώ εδώ. Πρωτού να ξαναδώσω το λόγο στη Συμπρόεδρο, θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις για να τονίσω τα όσα λέχθηκαν από τους δύο συνεισηγητές. Υπάρχει ένα πρόβλημα τύπου και μορφής, όπως υπενθύμησε ο κύριος Δεγκράντες Πασκουάλ, διότι τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση άνευ προηγουμένου, διότι δεν ξέρουμε εάν οι δύο επιτροπές και οι συγητές θα πρέπει να εργαστούν πάνω στο κείμενο που παρουσιάστηκε, αν υπάρχουν συμπληρωματικές σημειώσεις της Επιτροπής, ποια από τις δύο επιτροπές μας θα ασχοληθεί με αυτά. Είναι κάτι το οποίο είναι τελείω νέο. Ε, ίσως μπορούμε να έχουμε εξηγήσει και η δεύτερη παρατηρήση που θέλω να κάνω είναι ότι υπάρχει, είναι κατεπίγους ανάγκη σχετικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει έναν κανονισμό που να επιτρέπει να παρουσιάσουμε ε, κάτι ε, που να έχουμε να αντιπαραθέσουμε απέναντι στις παγκόσμιες συμμαχίες. Έχουμε το πρόβλημα ε, της συζήτησης με τις Ηνωμένε Πολιτείε και είναι δύσκολο να συζητήσουμε με τις Ηνωμένε Πολιτείε για μέτρα ασφαλείας, ενώ τώρα ε, δεν υπάρχει καμία δράση, κανένας γενικός έλεγχος, ε, καμία πιστοποίηση για τα συστήματα εξοπλισμού ελέγχου αερομεταφορών των κρατών. Η Παγκόσμια Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Ηνωμένες πολιτείες ε, για την συμφωνία που υπάρχει ε, που μπορεί να απειλείται από προβλήματα ασφαλείας και αυτό είναι μια πραγματική δυσκολία για να συζητήσουμε ένα σύνολο συνεκτικό για τα μέτρα ασφαλείας με τις Ηνωμένε Πολιτείες και ίσως αύριο με άλλες χώρες ή ομάδες χωρών. Η σημερινή κατάσταση για τις ειδικέ συζητήσεις ασφαλείας με, ορισμένες, ε, με ορισμένα αεροσκάφη ε, μας δείχνει τη δυσκολία που έχουμε στη συζήτηση. Κυρία Συμπρόεδρε, σας δίνω τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα, έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις ε, για, και για τους δύο εισηγητές, αλλά θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο στην Επιτροπή για να έχουμε μερικές πρώτες απαντήσεις και θα ήθελα να δώσω τον λόγο στην κυρία Ναμπάλα Κάργο εκεί εφόσον έχουμε μόνο αυτόν τον περιορισμένο χρόνο αν θα μπορούσατε ε, σύντομα ε, να μας μιλήσετε. Επιτροπή έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα να λάβω τον λόγο σε αυτή τη μεικτή συνεδρίαση C-TRANS και ΙΜΚΟ και ε, στην ευχαρίστω ε, την εισηγη, τους εισηγητές. Έχω σημειώσει τις ερωτήσεις που τέθηκαν και ναι, σχετικά να ασχοληθώ με το περιεχόμενο ή με την κατάσταση την οποία υπάρχει. Θα αρχίσω με το περιεχόμενο και ε, να δούμε το στόχο της πρότασης. Μερικά σημεία τονίστηκαν από τον εισηγητή The Grandes Pasquale και η πρόταση έχει ως στόχο και είναι αρκετά δομημένη να εξασφαλίσει την ελεύθερη ε, κυκλοφορία των αεροσκαφών της πολιτικής αεροπορίας στις αγορές μας ε, σε σχέση επίσης με τους κλάδους τους οικονομικούς, τους ευρωπαϊκούς και να εναρμονίσουμε τα επίπεδα ε, στα αεροδρόμια. Η 3-2008 σχετικά με την ασφάλεια για την πολιτική αεροπορία έχει προδιαγραφές τεχνικές ε, και επίσης απαιτήσει ε, επιδόσεων. Αλλά αυτή η νομοθεσία, όπως, είπε, όπως λέχθηκε, δεν συμπληρώνεται από ένα νομικό σύστημα δεσμευτικό ε, και ένα πιστοποιητικό για να εξασφαλιστεί ότι τα επίπεδα, τα πρότυπα που απαιτούνται όντως πληρούνται στην πραγματικότητα. Σχετικά με το στοιχείο, το βασικό της πρότασης, δηλαδή να υπάρξει ένα σύστημα πιστοποίησης δεσμευτικό για κάθε τύπο αεροσκάφους που να υπάρχει να τίθεται σε διάθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει της αρχής ε, της αμοιβαία αναγνώρισης τροπολογία 10 που δεν υπάρχει για την ώρα. Δεύτερον, η χρήση ε, μια κοινή μεθοδολογία ελέγχου και κοινή μεθόδου πιστοποίηση του εξοπλισμού που δεν υπάρχουν για την ώρα. Ε, με τρόπο νομικά δεσμευτικό. Τρίτον, ε, στις ε, διορισμένα όργανα να εγκρίνουν τη συμμόρφωση το, του εξοπλισμού με τις απαιτήσει αποδόσεως που βάσει της επιστοποίησης του τύπου έγκρισης, της έγκρισης τύπου και επίσης η υποχρέωση των κατασκευαστών όταν τοποθετούν τον εξοπλισμό αυτό στην αγορά ε, να, ε, να λάβουν υπόψη το πιστοποιητικό συμμόρφωσης βάσει του του, της, της νέας έγκρισης τύπου. Ο εισηγητής είπε ότι το προτινόμενο σύστημα βασίζεται στην διάσκεψη στην ΕΚΑΚ που αναπτύχθηκε από τα κράτη-μέλη ε, για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του εξοπλισμού βάσει των απαιτήσεων. Και ε, υπάρχει μια κοινή μεθοδολογία ελέγχων, ένα σύστημα για την έγκριση του ελεγχόμενου εξοπλισμού, αλλά που δεν είναι κάτι το νομικά δεσμευτικό. Η πρόταση συνδυάζει το σύστημα αυτή με μία ε, διαδικασία εξουσιοδότησης, έγκρισης σχετικά με τα εργαστήρια κλπ. Σήμερα δεν υπάρχει υποχρέωση δεσμευτική για τον κατασκευαστή να συμμορφούται με την κοινή αξιολόγηση της ΕΚΑΚ. Ε, το σύστημα, τα συστήματα πιστοποίησης των κρατών μελών διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ο εξοπλισμός που πιστοποιείται σε μια χώρα έχει μόνο μια εγγύηση ε, μόνο σε αυτήν την χώρα. Ε, ο κατασκευαστής εξοπλισμού πρέπει να περάσει από διάφορες διαδικασίες πιστοποίησης αν θέλει σε πάρα πολλές χώρες να θέσει στην αγορά τον εξοπλισμό του. Ο κανονισμός θα ήθελε να τα διορθώσει όλα αυτά ούτως ώστε το σύστημα της ΕΚΑΚ να είναι νομικά δεσμευτικό να υπάρχει μια σήμανση ε, σχετικά με το πιστοποιητικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα σημαντικό θέμα που θέτουν οι ενδιαφερόμενοι είναι ότι με την ε, νομικά δεσμευτική φύση αυτό σημαίνει ότι όλοι οι διαγωνισμοί, όλες οι δημόσιες συμβάσεις ε, για εξοπλισμό από στα αεροδρόμια απαιτεί ένα νέο, μια νέα έγκριση τύπου. Υπάρξουν διαφορές στις χώρες μέλη σχετικά με αυτό που ζητούν για τις προσφορές σε διαγωνισμούς για την παροχή αυτού του τύπου εξοπλισμού. Υπάρχει εδώ ένα θέμα ασφαλείας. Τώρα τα, οι δυσκολίες που αναφέρθηκαν από τους εισηγητές ε, και τον πρόεδρο ε, θα πρέπει να υπάρχει μια θετική μέθοδος όλα τα ε, μέλη να, μαζί να συμφωνήσουν. Υπάρχει μια συζήτηση με τις Ηνωμένε Πολιτείε σχετικά με τις συσκευές της ηλεκτρονικές και να υπάρξει εμπιστοσύνη επίσης με τους διεθνείς εταίρους μας που μπορούν ε, να είναι ε, διασφαλισμένοι ότι έχουμε τον εξοπλισμό για την ανείχνευση εκρηκτικών. Σχετικά με τον κλάδο βεβαίως έχουμε έχουμε συμβολή των αντιπροσώπων του κλάδου λέγοντας ότι το σύστημα της ΕΚΑΚ για κοινή μεθοδολογία ε, λειτουργεί καλά, αλλά η έλλειψη ε, ενός ενιαίου πιστοποιητικού τους επηρεάζει όταν θέλουν ε, να τοποθετούν τον εξοπλισμό σε κάθε εθνική αγορά και σε ανταγωνισμό με άλλους εξοπλισμούς στους διαγωνισμούς. Αυτό λέχθηκε από την Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια που είναι ε, βασικός φορέας για την ασφάλεια. Επίσης η ΑΙΑΤΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση για την διοικητική επιμέλεια που έχουν, έχουν πιστοποιητικά μιας χρήσης και ε, επίσης ε, για τα φορτία γίνεται κάποιος έλεγχος. Ε, έχουν διαρρομεταφορές για, το, για τον έλεγχο, για το screening των φορτίων για κάθε χώρα και η διεθνής αναγνώριση του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται είναι κάτι το βασικό και ιδαλλιώς θα πρέπει να ελέγχουν ε, τα φορτία όταν ε, προσπαθούν να εισέλθουν σε χώρες όπως οι Ηνωμένε Πολιτείες. Και αυτό έφεραν στην προσοχή μας. Επίσης, το Διεθνώς Συμβούλιο Ξεγωγών και η ΚΑΟ ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό. Σχετικά με την κατάσταση των πραγμάτων, σημείωσα προσεκτικά τις ανησυχίες σχετικά με τη μορφή, την διαδικασία και ε, θα ασχοληθώ με τα γεγονότα. Η πρόταση που υιοθετήθηκε τον Σεπτέμβριο παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Συμβούλιο στις 22 Νοεμβρίου και δεν τοποθετήθηκε ε, στην ημερήσια διάταξη κάποιου Συμβουλίου από τότε. Νομίζουμε ότι τα συμπεράσματα είναι σημαντικά ε, και παραμένουν σε λανθάνουσα κατάσταση. Νομίζουμε ότι αυτή η πρόταση δεν ε, παραλήφθηκε κανονικά από τα κράτη-μέλη. Χρειάζεται χρόνος λοιπόν για να ξανασταθούμε στα πόδια μας και να κατανοήσουμε γιατί δεν υπήρξε προεδρία μέχρι τώρα που να επιθυμούσε να βάλει την πρόταση επιτάπητος. Δεν υπήρξε διάλογος με το Συμβούλιο σχετικά με την πρόταση αυτή εμείς κλεθήκαμε, εμείς η DigiHome, να παρουσιάσουμε την πρόταση στην ΕΚΑΚ, στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη της Πολιτικής Αεροπορίας, στους εμπειρογνώμενες της διοίκησης κληθήκαμε και ο υποδιευθυντής μας παρουσίασε την πρόταση στους Γενικούς Διευθυντές Πολιτικής Αεροπορίας στην συνεδρίαση που εξαμηνία που έχουν και κληθήκαμε πιο πρόσφατα να παρουσιάσουμε την πρόταση στους ε, ενδιαφερόμενους ομάδες ασφαλείας που εκπρόσωποι κατασκευαστών, εμπειρογνώμονες από κράτη-μέλη, σε αυτή την ομάδα αντιπροσωπεύονται όλοι αυτοί. Αυτή είναι η κατάσταση ως έχει σήμερα. Εμείς έχουμε εξετάσει ε, την κατάσταση στα ε, κράτη που ενδιαφέρονται περισσότερο και αυτό είναι κανονικό, είναι κανονική διαδικασία. Ε, συνεργαζόμαστε με τέσσερα ή πέντε κρατημέλη διμερώς για να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε ποιες είναι οι πραγματικές τους ανησυχίες και όπως αναφέρθηκε προηγουμένως οι ανησυχίες δεν ξέρουμε αν είναι πραγματικές ανησυχίες είναι τα επιχειρήματα και ότι από και πίσω υπάρχουν ε, ανησυχίες πιο σημαντικές. Πρέπει να κατανοήσουμε την κατάσταση. Ε, μία από τις ανησυχίες που εκφράστηκε, όπως λέχθηκε και προηγουμένως, είναι η αντίληψη ότι η Κομισιό ε, προτείνει ένα νέο σύστημα ε, να αντικαταστήσει το σύστημα ΕΚΑΚ με το οποίο αυτές οι πέντε ε, χώρες ήταν ικανοποιημένες και κρατος μέλος υποστηρίζει την ΕΚΑΚ σχετικά με τη νέα πιστοποίηση. Δεύτερον, επίσης μια άλλη ανησυχία σημαντική που μπορούμε να επαληθεύσουμε είναι ότι η πρόταση θα εμποδίσει τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν πιο αυστηρά μέτρα ε, μετά την, ε, τον κανονισμό του 2008. Δεν είναι η περίπτωση αυτή μια τέτοια πρόταση δεν θα επηρεάσει την νομική ισχύ ε, του κανονισμού 300 του 2008 και την δυνατότητα κρατών μελών να υιοθετούν πιο αυστηρά μέτρα. Ε, οι λόγοι είναι ότι δεν υπήρχε ε, δυνατότητα να παρουσιαστούν οι επιλογές. Δεύτερον, όπως αναφέρθηκε από τον κύριο Ντεγκράντες, είναι το άρθρο 4, το, τα κράτη-μέλη δεν θα επιβάλλουν επιπλέον απαιτήσει σε σχέση με το πιστοποιημένο εξοπλισμό. Αυτές οι πρόσθετες απαιτήσει δεν είναι τα πιο αυστηρά μέτρα. Έχουν σχέση με την διαδικασία πιστοποίησης αυτή καθεαυτή και όχι με τις απαιτήσει σχετικά με την ε, επίδοση. Ναι. Σας παρακαλώ γιατί έχουμε και ερωτήσεις. Λοιπόν, η συζήτηση θα πρέπει να μας επιτρέψει να αναγνωρίσουμε ποιες διατα... αν οι διατάξεις είναι χρήσιμες ή δεν είναι. Υπήρχε και το άρθρο 10 που οδήγησε στην ΑΔΕΑ ότι έχουμε, ότι προτείνονται νέα μέλη για την ΕΚΑΚ που δεν είναι η περίπτωση ε, σχετικά με την ανάγκη να υπάρχει μια αρχή ε, επίσης και συστητικά με ε, τον, τον φόρτο των επιπλέον που επιβάλλεται από τις πρόσθετες απαιτήσεις. Ε, ορισμένοι λένε ότι δεν εξετάζουμε αρκετά τα θέματα ασφαλείας και βασιζόμαστε στις ανάγκες της αγοράς. Η Κομισιόν τώρα προσπαθεί να ε, συνεργαστεί με τους δύο συνομοθέτες, με συνεδριάσεις, με τους συναδέλφους των δύο αρμοδίων επιτροπών εδώ και είναι χρήσιμη συνεδρία σήμερα. Προσπαθούμε να συνεργαστούμε με το Συμβούλιο και την Εστονική Προεδρία, ούτω ώστε να προχωρήσουμε σχετικά με το θέμα αυτό. Η Επιτροπή ευχαριστεί τον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την συνεργασία. Ευχαριστούμε. Εντάξει, πολύ σας ευχαριστούμε. Ως συνήθως είχαμε μια πρώτη παρουσίαση των προτάσεων και επειδή συμφωνήσαμε να είναι μεικτή συνεδρίαση θα δώσουμε το λόγο στους όντως εισηγητές και τα λοιπά μέλη που επιθυμούν να παρέμβουν και από τις δύο επιτροπές για να θέσουν ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Κουέλιου. Όχι, δεν θέλετε. Η κυρία Γκραπίνη λοιπόν. Συνεισηγήτρια. Ε, ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Πέραν των παρατηρήσεων καλά θα, των εισηγητών καλό θα ήταν να παρέμβουν και σκιώδεις για να έχει μια σφαιρική ε, εικόνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε και εμείς το δικό μας ρόλο εδώ, όχι μόνο οι καθήλυνα αρμόδιοι εισηγητές. Εγώ λοιπόν είμαι σκιώδης εισηγήτρια από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες από την Επιτροπή Τραν. Η συνάδελφος που είναι υπεύθυνη από την ΕΜΚΟ μου ζήτησε να μεταβιβάσω τις απόψεις της. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το συνολικό τοπίο της πρότασης, το σκηνικό εντός του οποίου υποβάλλεται το 2015 εγκρίθηκε η Ευρωπαϊκή Ατζέντα, το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Ασφάλεια. Και βάσει αυτού του θεματολογίου, ο κύριος Γιονκέρ υποστήριζε ότι πρέπει να υπάρξει μια ένωση για την ασφάλεια. Άρα ένας ενιαίος κανονισμός ήταν αυτό που χρειαζόταν. Ωραία. Ίσως έγιναν επικοινωνιακά σφάλματα από την πλευρά της Επιτροπής και όχι μόνο. Τέλος πάντων έχουμε βρεθεί και πάλι σε μια κατάσταση που υπάρχει διαφωνία. Κατά την άποψή μου είναι πολύ σημαντικό αυτό που έρχεται τώρα ως μήνυμα. Να μην χάσουμε άλλο χρόνο. Σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής μπορούμε να βελτιώσουμε το περιεχόμενό της. Όπως εξήγησε ήδη η Επιτροπή ως προς την μορφή και το περιεχόμενο. Ως προς τις επιφυλάξεις και τους ενδιασμούς των κρατών μελών. Μπορούμε να βελτιώσουμε την έκθεση και θα ήταν σημαντική απώλεια χρόνου εάν την αποσύραμε για να την ξαναποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει λοιπόν να εργαστούμε βάσει αυτής της πρότασης. Ο εισηγητής της ΤΡΑΝ θα οργανώσει συνομιλίε με όλου εμά για να το διαπραγματευτούμε. Άρα πρέπει να δουλέψουμε. Τι μετράει περισσότερο λοιπόν. Η ασφάλεια είναι σημαντική για όλους και κατά δεύτερον για αυτά τα συστήματα ασφαλείας οι δαπάνες είναι τεράστιες από την πλευρά των αρμόδιων φορέων και των εμπορευμένων. Θέλουμε ένα σύστημα αποτελεσματικό και ενίο για τον έλεγχο ασφαλείας και την πιστοποίηση των εξοπλισμών. Και δεν θέλουμε να αποκλείεται η δυνατότητα, να κράτος μέλος, αν θέλει, να έχει αυστηρότερους κανόνες. Όπως σωστά διευκρίνησε και η Επιτροπή. Όμως αυτή την ενιαία αγορά των 15 δις ευρώ, γιατί αυτή είναι η αξία των συσκευών screening, πρέπει να υπάρχει έστω αυτή η υποχρέωση, μια, ε, ενιαία, ε, ένα ενιαίο σύστημα έγκρισης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το άρθρο 31 προτείνει οι συσκευές screening να εγκρίνονται από τα κράτη-μέλη βάσει τυποποιημένων διαδικασιών και να αγοραστούν, να τοποθετηθούν στα αεροδρόμια πριν από τη λήξη του προηγούμενου κανονισμού για να υπάρξει συνέχεια και να εξασφαλιστεί περίοδος ε, χρήσης, μεταβατική περίοδος. Θα πρέπει όμως, εάν υπάρχει τέτοια συγκεκριμένη ημερομηνία, να λάβουμε υπόψη ότι θα είναι πολύ μεγάλες οι δαπάνες. Ε, τρία χρόνια μεταβατική περίοδος και μετά εγγύησει. Θα πρέπει λοιπόν να συμπληρώσουμε το άρθρο με κάτι, με ένα εδάφιο, μια παράγραφο, κάτι. Επίσης πρέπει να προβλέψουμε ορισμό για τις τεχνικές υπηρεσίες χωρίς ε, ρητή μνήμα. Στο άρθρο 8.2 ή 8.1 πρέπει να προσθεθεί μια διάταξη για τον αποχρωτικό χαρακτήρα ε, που θα έχει για τον παραγωγό να λάβει εξουσιοδότηση για τις συσκευέ screening. Και μετά το θέμα των ακτινοβολιών. Μην το ξεχνάμε, ε, είμαστε κι εμείς πολίτες, περνάμε από αυτές τις συσκευές screening και κανείς δεν μας λέει αν είμαστε προστατευμένοι ή όχι ως προς την ακτινοβολία των συσκευών. Η ομάδα μου λοιπόν θα υποβάλει σχετικά τροπολογίες, όμως επί της ουσίας θα ξεκινήσω από το σημείο από το οποίο ξεκίνησα. Δεν χρειάζεται να τα ξεκινήσουμε όλα από το μηδέν. Μπορούμε απλώ να βελτιώσουμε την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μεμονωμένα για συγκεκριμένα στοιχεία να ε, διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο και συγκεκριμένε χώρε. Οι μικρέ χώρε έτσι κι αλλιώ δεν έχουν πάντοτε την ε, δυνατότητα να κάνουν την άποψή του να βαρύνει. Οπότε στην ουσία θα έχουμε έναν κανονισμό που θα επιλύει το πρόβλημα τη ε, νέα πιστοποίηση στην εσωτερική αγορά διασφαλίζοντας την προστασία των πολιτών από την πλευρά της υγείας και της ασφάλειας με αυτού του είδους ενιαίας ε, ε, εξουσιοδότησης. Διότι πραγματικά τα έξοδα που γίνονται αυτή τη στιγμή στα αεροδρόμια για τις συσκευές είναι τεράστια. Δεν το αποφύγουμε αυτό. Ευχαριστώ. Μιλήσατε για δύο. Πραγματικά και κυριολεκτικά. Και επειδή μιλήσατε και για την κυρία Χέτ, ο λόγος στην κυρία Φώστερ για του συντηρητικού και μεταρρυθμιστές, οι οποίοι θα μιλήσει, η οποία θα μιλήσει εκ μέρου του κ. Βαντάλεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο σκιώδη μα ο Πέτρε Βαντάλεν, δεν είναι εδώ. Όμω, ήδη από την 11η Σεπτεμβρίου έχω ασχοληθεί με το θέμα των συσκευών ε, screening στα αεροδρόμια και το γνωρίζω πολύ καλά, εκτό που δούλευα και εγώ σε τέτοια εταιρεία αεροπορική. Να υπογραμμίσω λοιπόν ότι η ασφάλεια και η ασφάλεια στην αεροπλοεία είναι η ουσία της δουλειάς της ICAC. Δηλαδή η διάσκεψη της πολιτικής αεροπορίας της Ευρώπης. Έχει δημιουργηθεί πριν από 60 χρόνια και συμμετέχουν 24 χώρες. Είναι ο μόνος οργανισμός που παρακολουθεί την, ε, τις επιταγές της ΙΚΑΟ, του Διεθνούς Αντίστοιχου Οργανισμού. Και η δουλειά τους είναι ακριβώς να τα συνδυάζουν όσα προκύπτουν από τη μια. Ακόμα και για την ασφάλεια στα αεροδρόμια τώρα, όλες οι αναφορές για τη συμμόρφωση την οποία επιδιώκουμε προκύπτουν από την ΙΚΑΚ.30 που ονομάζουμε. Αυτή είναι, αυτό είναι το σύνολο των κανόνων που ισχύει τώρα. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής λοιπόν, Επιτροπής κατά πρώτον παραβιάζει την αρχή των πρωτοκόλων επικουρικότητας, το πρωτόκολλο 2 του άρθρου 6, διότι εδώ τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα. Δεν λέω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν λόγο να ενδιαφέρονται και μάλιστα ενεργά ε, και να συμμετέχουν στι όλε τι διαπραγματεύσει. Αλλά ένα-δυο σημεία από την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μόνο να κοιτάξει κανεί. Δεν λαμβάνονται υπόψη όσο έχουν γίνει για την ευελιξία που απαιτείται λόγου χάρη για τα περισσότερα αυστηρά μέτρα. Κάποια κρατημελή τα χρειάζονται. Διότι ε, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερε απειλέ από άλλου, από την τρομοκρατία λόγου χάρη. Επίση, η διαδικασία αξιολόγηση ε, είναι λιγότερο αυστηρή βάση. Δημιουργούνται διπλά μέτρα και σταθμά κάπω. Η Αυστραλία, ο Καναδά, οι ΗΠΑ, το Ισραήλ έχουν αυστηρά μέτρα. Εδώ λοιπόν χρειάζονται τεράστιε προσπάθειε συνεννόηση ε, μυστικών υπηρεσιών και οι πληροφορίε που ανταλλάσσουμε μεταξύ μα είναι πολλέ ε, και σημαντικέ. Επίση, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προκυπλέψουν αυτά τα αυστηρότερα μέτρα όταν έχουν ε, σημαντικότερε ανάγκε. Εδώ λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιουργεί κίνδυνο έκθεση ευαίσθητων πληροφοριών, επίση αύξηση γραφειοκρατία και επιπλέον κόστο που δεν χρειάζονται. Και εγώ προσωπικώ θα πρότεινα απλώ το status quo να υπερισχύσει. Δεν λέω ότι μπορεί να μην χρειαστούν ε, κάποιε προβλέψει στο, μέλλον. Όμω, να σα πω ότι εγώ είμαι διαρκώ επαφή με εταιρείε ασφαλεία. Δεν είχα ποτέ καμία συνομιλία ή συνάντηση με κάποιον που να ασχολείται με εξοπλισμό ασφαλεία από αυτό το χώρο και του ανθρώπου που εργάζονται εκεί που να είχε πρόβλημα με το status quo και τον τρόπο που αντιμετωπίζει το όλο θέμα η ICAC. Η ICAC. E ε, ε, εδώ λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να τα λάβει αυτά υπόψη. Ε, για αυτού του βασικού λόγου, θα υπάρχουν προφανώ και άλλοι και μπορούμε να του συζητήσουμε από μακρόν, πιστεύω η πρόταση αυτή μπορεί να αποσυρθεί. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε να προτείνει κάτι καινούργιο στο μέλλον, ε, δεν είναι ένα θέμα σήματο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ούτω καθεξή. Έτσι κι αλλιώ η ΕΚΑΚ θα κάνει όλε τι δοκιμέ, όλα τα τεστ, δεν θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπότε δεν υπάρχει καμία απέτηση να αλλάξουν τα πράγματα σε σχέση με αυτό που γίνεται τώρα. Ο κανονισμός ε, δεν χρειάζεται καν. Μια οδηγία θα ήταν πιο εύστοχη. Αυτό θα έλεγα στου συναδέλφου, διότι τα κράτη-μέλη πρέπει απλώ να διατηρήσουν την ευελιξία σε αυτή τη δράση και ε, το ίδιο και το Κοινοβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν ήθελα να κάνω αυτά τα σχόλια και νομίζω ήταν σημαντικό να έχουμε αυτή την ακρόαση και σα ευχαριστώ θερμά που την οργανώσατε, διότι όσο ακούσαμε ω τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφήνουν ε, πολλέ από τι προσδοκίε μα ε, ανικανοποιητέ. Και νομίζω είναι πολλά αυτά που μπορούμε να κάνουμε, αλλά στο μέλλον δεν είναι αυτό ο τομέα στον οποίο χρειάζεται τώρα να παρέμβει η Επιτροπή, υπάρχουν πολλοί άλλοι. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Η ε, κυρία Χουισμένοβα από τους Φιλελευθέρους και όλες εισηγήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της Eurostat από το 2015, ο συνολικός αριθμός των ταξιδιωτών που χρησιμοποιούν την αεροπλοεία ετησίως στην Ευρώπη είναι περίπου 218 εκατομμύρια. Εκατοντάδες χιλιάδες άτομα ταξιδεύουν για λόγους ε, δουλειάς, αυθημερών, και αυτό επιβάλλει να βρούμε μια λύση ισόρροπη και εξυγχρονισμένη για τον τομέα της αεροπλοείας, όπου ο κατακαιρματισμός των δοκιμών, διαφορετικά, τα διαφορετικά συστήματα πιστοποίησης δημιουργούν, δημιουργούν δυσκολίες στις εγκαταστάσεις των αεροδρομίων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να καλύψει τις διαφορές των απαιτήσεων και των προτύπων και την μεθοδολογία των δοκιμών και της πιστοποίησης των εξοπλισμών ασφαλείας στα αεροδρόμια. Ε, κατά τρόπο ώστε ο κατακαιρματισμός της ενιαίας αγοράς να διορθωθεί, επιτρέποντας οι εξοπλισμοί που πιστοποιούνται σε ένα κατός μέλος να πιστοποιούνται ταυτόχρονα και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να μειώσει το κόστος και τους φραγμούς, τους ρυθμιστικούς φραγμούς και να δημιουργήσει θετική μόχλευση για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εταιριών. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν έχω δύο ερωτήσεις για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρώτη είναι ε, σύμφωνα με την ΕΟΚΕ, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η έγκριση της εξοδότησης των εξοπλισμών από μία Ευρωπαϊκή Αρχή θα είναι αποτελεσματικότερη, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προβλέπει τη δημιουργία τέτοια αρχή. Γιατί και η δεύτερη είναι τι να κάνουμε για την επικουρικότητα. Η πρόταση μεταφέρει εν μέρη εθνικέ αρμοδιότητε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μου δώσει μια απάντηση πιο συγκεκριμένη για την πρόοδο που έχει επιτελεστεί για να βρούμε μια κοινή θέση στο Συμβούλιο για τη δημιουργία ενός ε, συστήματος ε, ευρωπαϊκής πιστοποίησης των εξοπλισμών ασφαλείας που χρησιμοποιούνται στα αεροδρόμια. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Εάν δεν υπάρχουν άλλες ή κάποιοι που θέλουν να μιλήσουν εκ μέρους του. Δεν βλέπω κάποιον άλλο συνάδελφο να θέλει το λόγο, οπότε να δώσω πάλι ε, το μικρόφωνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει στο λίγο χρόνο που μας έχει μείνει στις ερωτήσεις που τέθηκαν στα σχόλια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Σε σχέση με το άρθρο 30 και την ανάγκη να ξαναδούμε τον κατάλογο για τη μελέτη δικτύπου, χρειάστηκε να προβλέψουμε μια περίοδο αρκετά ε, άνετη για τα κράτη-μέλη. Η πρόταση που γίνεται, που έγινε μάλλον, την σημειώνουμε για να εξετάσουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε καλύτερα το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 30. Ως προς τις πτυχές safety, ασφάλεια. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο καλύπτεται στο άρθρο 9 και 17 της πρότασης. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, ε, οι κίνδυνοι που δημιουργούνται και προκαλούνται από τον εξοπλισμό και οποιαδήποτε πρόταση σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις της ακτινοβολίας και το καθεξής, είναι στοιχεία που τα κοιτάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ευχαρίστως να τα λάβει υπόψη για να διασφαλίσει ότι η ασφάλεια και η προστασία συμβαδίζουν. Ως προς τις παρατηρήσεις για την ΕΚΑΚ. Α, θα συμφωνήσουμε απολύτως. Η ΕΚΑΚ είναι ένα σύστημα ε, εύρωστο. Έχει εξελιχθεί πολύ θετικά και έχει πολύ καλές επιδόσεις. Έχει πολύ καλές επιδόσεις στα πλαίσια της εντολής της με μια πολύ καλή μεθοδολογία. Όμως όπως εξήγησα στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις, δεν ε, έχει νομικώς δεσμευτική αξία και στην προσοχή μας έχουν υποπέσει περιπτώσεις εξοπλισμού που δεν πέρασαν τις δοκιμές της ΕΚΑΚ και μετά τέθηκαν στην αγορά και έφτασαν στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Αυτό μας το εντόπισε η ίδια η ΕΚΑΚ. Δεν υπάρχει νομική κοινωνική υποχρέωση. Οπότε δεν είναι προϋπόθεση σε μια δημόσια προμήθεια η έγκριση της ΕΚΑΤ για να τοποθετηθεί κάτι στα αεροδρόμια. Ε, Ω προ τα αυστηρότερα μέτρα, υπογραμμίζω ξανά, ο κανονισμός 300 του 2008 συνεχίζει να ισχύει. Δεν επηρεάζεται το δικαίωμα των κρατών μελών βάσει του κανονισμού αυτού. Οποιαδήποτε διατύπωση, ακόμη και αν είναι νομικός περιττή, Εάν χρειάζεται για σαφήνεια, ας υπάρχει στο αναθεωρημένο κείμενο, ε, γιατί προφανώς έλειπε. Ως προς την ε, άποψη της ΕΟΚΕ και την επιλογή να υπάρχει μια ενιαία αρχή, ευρωπαϊκή αρχή, αυτή ήταν μια από τις εναλλακτικές που μελετήσαμε στη μελέτη αντικτύπου και ε, απορρίφθηκε, απορρίφθηκε διότι θεωρήσαμε ότι σε σχέση με, την, ε, με τις απαιτήσει που θα προκαλούσε και την τάση της Επιτροπής να αποφεύγει να δημιουργεί νέους οργανισμούς και να τους επανδρώνει έτσι το αναλύσαμε και η επιλογή αυτή ε, απορρίφθηκε. Απέναντίας η ΕΚΑΚ υπάρχει, κάνει φοβερή δουλειά, οπότε από την άποψη ε, σωστής διαχείρισης των πόρων ήταν η καλύτερη επιλογή το πιστοποιητικό να ισχύει πέραν των όσων γίνονται ούτως ή άλλως επιτυχώς από την ΕΚΑΚ. Ελπίζω ότι απήντησα στις ερωτήσεις και εάν υπάρχουν ακόμα πιο συγκεκριμένα ερωτήματα, ευχαρίστως να τα παραλάβουμε για να τα απαντήσουμε γραπτός. Θα επαναλάβω ότι παραμένουμε στη διάθεσή σας για να βοηθήσουμε το Κοινοβούλιο και τις δύο επιτροπές σας να μελετήσουν το θέμα αυτό. Ε, Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή για τις ε, πληροφορίες αυτές. Εγώ δεν έχω άλλα ε, σχόλια, αλλά θα δώσω τον λόγο στον συνηγητή από την Επιτροπή Τραν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και συνεισηγητρία. Στην Επιτροπή Μεταφορών εδώ και πολλά χρόνια εργαζόμαστε στη συναπόφαση και ξέρουμε ότι πολλές φορές χρειάζεται να αλλάξουν οι διαπραγματεύσεις. Αυτά όλα είναι άσκοπα και μάταια, διότι κοφεύει το Συμβούλιο ή μας αγνοεί. Για να μην ε, χάνει χρόνο, ε, για να ασχολείται με πράγματα άσκοπα και εμείς πολλές φορές χρειάζεται να ανακρούσουμε πρίμνα για να έχει νόημα η δουλειά μας. Η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής χωράει βελτίωση από το Κοινοβούλιο, χωράει, αλλά να μην είναι μάταια η δουλειά μα γιατί και η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή ομολογεί πραγματικά ότι είμαστε σε ένα πολιτικό κενό, είμαστε μετέωροι. Το Συμβούλιο έβγαλε ένα φιρμάνι και αγνοεί τους υπολείπους. Ωραία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει τις δυσκολίες και λοιπόν Μπορεί να είναι εύλογο όλα αυτά, αλλά και η κυρία Φώστερ, την οποία σέβομαι και τιμώ, ε, επικαλείται την επικουρικότητα. Και τα ξέρει αυτά και ο κύριος Κοέγιο που δουλεύει πάρα πολύ στην Επιτροπή Ελευθεριών. Η ασφάλεια είναι θέμα ε, κρατικής αρμοδιότητας. Αλλά σήμερα προσπαθούμε να τα ξεπεράσουμε αυτά για να καλύψουμε τις ανάγκες που έχουν αλλάξει σήμερα ως προς την ασφάλεια. Θέλω να σας πω το εξή. Ο ίδιος ο πρόεδρος Γιούνκερ μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις Βρυξέλλες στις 23 Μαρτίου πέρσι είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια ένωση ασφάλειας για να αντιμετωπίσει την ε, τρομοκρατία αποτελεσματικά και στις 20 Απριλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια πρωτοβουλία. Άρα ε, τώρα θα πρέπει να λύσουμε αυτά τα θέματα. Αυτό πώς λύνεται, με τους εξής δύο τρόπους. Πρώτον, είτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει αυτή την αρμοδιότητα, την πρωτοβουλία, θα αποσύρει και θα φέρει νέα πρόταση, ε, σύμφωνα με τα όσα είπε το Συμβούλιο, κάτι πιο βιώσιμο, εν πάση περιπτώσει, που εγώ προτείνω αυτό, αυτό είναι το ένα, ή το δεύτερο, να φέρει ένα ε, συμπληρωματικό, διορθωτικό μνημόνιο, κάτι που να λέει ε, ότι αλλάζω αυτά που ήταν ε, απαράδεκτα, εν πάση για να προχωρήσει η πρόταση. Όλα τα υπόλοιπα είναι φιλολογίες. Αυτά είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα τα επιχειρήματα είναι σεβαστά και όλε οι απόψει. Αλλά τώρα, για να είμαι ειλικρινή, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δεχτεί τα όσα προτείνει το Συμβούλιο, δεν θα προχωρήσει το Συμβούλιο, δεν είναι βιωσιμότητα σε αυτή την υπόθεση. Και ξέρετε, άλλο είναι η αρμοδιότητα των κρατών για την ασφάλεια που επικαλούνται την επικορικότητα και άλλο είναι να απαγορεύσουν την εναρμόνιση. Εδώ δεν απαγορεύεται η εναρμόνιση. Φαίνεται αδικαιολόγητο και ανεξήγητο αυτό το πράγμα. Και συγχώρητο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ειλικρινή. Λέει, ομολογεί ότι έχει δυσκολίε. Εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι να κάνει σε αυτό το κάδρο θα δουλεύουμε στο βρόντο. Για ποιο λόγο. Σέβομαι όλες τις απόψεις. Κατανοώ ότι η Κομισιόν δεν θέλει να απαντήσει την ερώτησή μου. Προτιμάει να το σκεφτεί αυτό που άκουσε και να μην δεσμευτεί τώρα. Ε, κάποια στιγμή να μας πει όμως τι θέλει. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θέλω να δώσω το λόγο τώρα στον Σύμπροεδρο μου, παρακαλώ. Euh. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα απλώς ε, να πω κάποια συμπεράσματα σε σχέση με τα όσα ακούσαμε. Μπορεί κανείς να σκεφτεί ως προς την ουσία υπάρχει ενδιαφέρον και συμφέρον να έχουμε πιστοποίηση και για λόγους ασφαλείας και για λόγους βιομηχανικούς και οικονομικούς, αλλά ότι υπάρχουν δυσκολίες επειδή αυτή η πρόταση της Κομισιόν είναι κατά κάποιο τρόπο ε, σε κατάσταση λίθαργο στο Συμβούλιο. Μπορεί, πρέπει να ζητήσουμε από την Κομισιό να αναφερθεί στις, ε, στο Προεδρείο των δύο Επιτροπών και να μας πει σαφώς ότι πρώτον διατηρεί τη θέση της όσα ε, έχει με τροποποίησεις και ότι αυτή η πρόταση με ή χωρίς προστίκη έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο για να ξαναεισέλθει μέσα στη διαδικασία συναπόφασης. Δηλαδή ε, να μπει στο στόχαστρο. Βεβαίως ε, αυτοί οι συνεισηγητές ε, δεν εργάστηκαν για το τίποτα για αυτόν τον φάκελο που παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση. Έχουμε διμερείς ε, σχέσεις, διμερείς επαφές ε, με ορισμένα ε, κράτη, τα οποία έχουν επιφυλακτικότητα και ως προς την επικουρικότητα επίσης η Κομισιό μπορεί να μας γράψει, να μας γράψει λέω, να μας γράψει και να μας πει ότι επαναδραστηριοποιείται αυτός ο φάκελος με την συμφωνία του Συμβουλίου ε, για διαδικασία συναπόφασης όσο έχει ή με προσθήκες, αντέντα, για να ξέρουμε ε, γιατί εργάζονται και για ποια στιγμή, για ποιο χρόνο θα μπορεί η Κομισιόν να μας γράψει προς τη μία ή άλλη κατεύθυνση, διότι αυτός ο φάκελος δεν μπορεί ε, να θεωρηθεί ότι έχει κάπως εξεταστεί, θα πρέπει να υπάρχει επαναδραστηριοποίηση και ίσως ένα αντέντουμ για να δούμε με την ε, Κομισιόν και τους εισηγητές, ούτω ώστε η εργασία του Κοινοβουλίου να λάβει χώρα μέσα σε ένα επιχειρησιακό πλαίσιο που να είναι ασφαλές, διότι τώρα δεν υπάρχει βεβαιότητα, υπάρχουν αμφιβολίες. Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ με την πρόταση του Συμπροέδρου. Επίσης θα ήθελα να προτείνω επίσης να ενημερώστε την, την Προεδρία για την κατάσταση των πραγμάτων, ε, την Προεδρία που έχουμε τώρα και νομίζω ότι θα πρέπει οι συγητές ε, να συνεργαστούν μαζί για να δουν ε, τι θέση θα πρέπει να υιοθετήσουμε και θα ενημερώσουμε όλα τα άλλα ενδιαφερόμενα μέλη για τα επόμενα βήματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω άλλη μια φορά την Κομισιόν που ήρθε εδώ να μας ενημερώσει. Νομίζω ότι οι γραμματείες των δύο ε, επιτροπών θα έρθουν σε επαφή μαζί σας. Θα ήθελα να ευχαριστώ τα μέλη της ΣΥΜΚΟ και της ΤΡΑΝ που ήρθανε σε αυτή την συνεδρίαση και εμείς θα συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας στα πλαίσια της ΣΥΜΚΟ. Κρύβει